ο κύριος Πέντρο Σίλβα Περέιρα διορίζεται ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Υπάρχουν ενστάσεις? Όχι. Επομένως εγκρίνεται ο διορισμός του.